Τώρα θα έρθουμε στις αλλαγές καθώς και στην έγκριση μερίσια διάταξη. Για την σημερινή μερίσια διάταξη δεν έχουν υποβληθεί καθόλου αιτήματα αλλαγή. Για την Τρίτη είχε προβλεφθεί ότι αύριο θα συζητήσουμε την έκθεση του κυρίου Ίγκορ Σόλτες για το διορισμό ενός μέλους από την ε, Μάλτα στο ελεγκτικό συνέδριο. Ωστόσο, η ακρόαση του υποψηφίου θα πρέπει να αναβληθεί, γιατί δεν είναι δυνατόν ε, ε, να διεξαχθεί αυτή τη στιγμή. Η ε, προθεσμία των δύο μηνών, η οποία προβλέπεται από το κανονισμό 121.3, παρατείνεται συνεπώς. Η Γκουε ε, ζήτησε, καθώς και οι σοσιαλιστές, αλλά πρώτη η Γκουε, ε, ζήτησε μία δήλωση του Συμβουλίου και της ε, Επιτροπής σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία και τον αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα ε, και να συμπεριληφθεί ως πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη της Τετάρτης. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη και ως αιτιολόγηση ζήτησε η κυρία Σπινέλη το λόγο. Όπω ήδη αποφασίστηκε στη διάσκεψη των Προεδρών, ζητώ εξ ονόματο της πολιτικής μου ομάδα να συζητήσουμε την Τρίτη ένα δεύτερο ψήφισμα για τα ε, κράτος δικαίου στην Πολωνία, διότι εντωμεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εξέφρασε την ανησυχία της για το κράτος δικαίου, ε, όπως επίσης και η Επιτροπή της Βενετίας διότι το συνταγματικό δικαστήριο έχει παραλύσει, διότι υπάρχει μια διαδικασία έγκρισης νέας νομοθεσίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, παρακολούθηση των μέσων ενημέρωσης και του διαδικτύου και της αμβλώσης. υπάρχει λοιπόν, λοιπόν ανάγκη να συζητηθεί ένα δεύτερο ψήφισμα για την ε, νομιμότητά τους βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου. Νομίζω ότι η δημοκρατία μετά το Brexit είναι το πρώτο αγαθό το οποίο πρέπει να υπερασπιστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αναφέρομαι και στους τρεις ε, πυλώνες της συνταγματικής δημοκρατίας, ε, το καθολικό δικαίωμα ψήφου, αλλά και το κράτος δικαίου και τον διαχωρισμό των εξουσιών. Δεν ε, είναι παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα ενός κράτους μέλους, αλλά είναι μια έκκληση για αρχές ε, και κοινού νόμους, τους οποίους έχουμε προσυπογράψει όλοι υπογράφοντας τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 2 και 6. Εάν η πολωνική κυβέρνηση ή οποιαδήποτε άλλη μελλοντική κυβέρνηση ή παρούσα κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα η Ουγγαρία ή ε, ε, έχουμε και τα πρόσφατα προεδρικά αποτελέσματα στην Αυστρία, ε, θεωρούν ότι οι αρχές αυτές παραβιάζουν την ε, κυριαρχία τους, θα πρέπει να συζητηθεί όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα εκ νέου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σπινέλη. Τώρα ο κύριος Γκερέρο έχει το λόγο υπέρ της πρότασης ψηφίσματος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Στις αρχές της χρονιάς, στις 19 Ιανουαρίου πιο συγκεκριμένα, συζητήσαμε εδώ στο σώμα αυτό για την κατάσταση στην Πολωνία και μάλιστα την παρουσία της Πρωθυπουργού της Πολωνίας. Και οι περισσότεροι εδώ εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις, για κάποιες συνταγματικές παραβιάσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο κράτος αυτό και σύμφωνα με πολλούς οι παρεμβίες αυτές είναι ασύμβατες και με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις βασικές και θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στηρίξαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προχωρήσει σε διάλογο με την κυβέρνηση της Πολωνίας προκειμένου να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία, στο σεβασμό των αξιών καρχών αυτών. Την πρώτη προηγούμενου μήνα υιοθετήθηκε γνωμοδότηση εκφράζοντας την ανησυχία μας επειδή ακριβώ δεν είχε γίνει τίποτα, αντίθετα είχε παρεύει η κυβέρνηση στον ορισμό των ε, μελών του, ελεκτικού, του συνταγματικού δικαστηρίου, το οποίο κανονικά είναι το αρμόδιο για τη συνταγματική νομιμότητα στη χώρα αυτή. Αυτό και άλλα πράγματα απασχολούσαν την εποχή εκείνη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά αποτελούν αρκετούς λόγους νομίζω τόσους μήνες μετά να εκτιμήσουμε και πάλι την κατάσταση και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει την αξιολόγηση της σημερινής κατάστασης. Και στη Λίμπε τις προηγούμενες εβδομάδες υπήρξε ένα ψήφισμα που εγκρίθηκε από πολλές πολιτικές ομάδες, μεταξύ άλλων και ομάδων που στη διάσκεψη των Πρόεδρων αρνήθηκαν να μπει αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Οπότε, η θέση της δικιάς μου ομάδας είναι να συμπεριληφθεί την Τρίτη στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ πολύ. Κατά το ψηφίσματο, ο κύριο Τσερνέτσκι θέλει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ. Με εκπλήσει το αίτημα αυτό, όπως επίσης και η αιτιολόγησή του. Την προηγούμενη εβδομάδα η διάσκεψη των Προέδρων είπε ότι δεν θα υπάρξει συζήτηση για το ζήτημα αυτό και ήσασταν κι εσείς παρόν στη διάσκεψη αυτή των Προέδρων. Υπογραμμίζω ότι στην Πολωνία δεν συμβαίνει τίποτα που να δικαιολογεί μια νέα, επαναλαμβάνω, μια νέα συζήτηση για την κατάσταση στην Πολωνία. Έγινε πρόσφατα τέτοια συζήτηση εδώ. Συνεπώς, πιστεύω ότι το να επιβάλλουμε τη συζήτηση αυτού του θέματος τώρα δεν είναι καλό. Οι Πολωνοί το αντιλαμβάνονται σαν ανάμειξη στα ζητήματα της χώρας τους. Καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια συζήτηση θα έχει ε, αρνητικές επιπτώσεις και όχι θετικές. Πρέπει λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Τίμερμανς, πρώτο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος είπε ότι η Πολωνία θα διευθετήσει τα ζητήματά τη. Γίνονται συνομιλίες ανάμεσα στις πολωνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Οπότε το να επιβάλλουμε μια τέτοια συζήτηση, το να στηρίξουμε μια τέτοια πρόταση και μάλιστα αμέσω μετά το Brexit, μια πρόταση σαν και αυτή που μόλις κάνατε, είναι κάτι που το αντιλαμβάνομαι σαν ανάμειξη στα εσωτερικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή στις εσωτερικές υποθέσει της Πολωνίας και μάλιστα μετά από τόσα έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο σα ζητάω να μην στηρίξετε το αίτημα αυτό. Δεν πρέπει να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά σε μια χώρα τόσο σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον κανονισμό. Διαδικαστικό. Έχω να κάνω μία πρόταση, λέει ο κύριος Φεχώστατ. Γιατί είναι πολύ εύκολο να πούμε έγινε Brexit οπότε α, να μην μιλήσουμε για την Πολωνία. Ε, εντάξει, ας πάμε σπίτια μας τότε. Να μην μιλήσουμε για τίποτα πια εδώ. Είναι αναγκαίο, πρέπει να μιλήσουμε για την Πολωνία. Την κατάλληλη στιγμή βέβαια οι διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνουν χώρα. Βρισκόμαστε στη μέση της διαδικασίας. Οπότε, όπως το έχω πει και στους σοσιαλιστές συναδέρφους και εκείνους από την ΚΟΥΕ και από τους πράσινου να αποφασίσουμε σήμερα να συμπεριληφθεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη του Σεπτεμβρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει ολοκληρώσει το δικό της το έργο. Εμείς έχουμε ήδη ψηφίσει ψήφισμα. Ε, λοιπόν, τώρα να αποφασίσουμε ότι θα μπει στην ημερήσια διάταξη του Σεπτεμβρίου η συζήτηση αυτή. Να μην κάνουμε τίποτα στα βιαστικά, συμφωνώ, και η φωνή μας να ακουστεί τότε στην Πολωνία. Ευχαριστώ. Ναι. Αυτή είναι μια άλλη πρόταση η πάει ακόμα πιο μακριά. Αυτό δεν είναι απλό από την οπτική του κανονισμού, γιατί για το, για το Σεπτέμβριο δεν είναι δυνατόν. Θα πρέπει να η δική σας πρόταση να διαμορφωθεί έτσι ούτως ώστε να καλέσουμε την ε, Ολομέλεια να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη αυτή την ε, πρόταση. Έτσι θα πρέπει να γίνει διαδικαστικά. Ε, δεν ξέρω, θα πρέπει να ρωτήσουμε τους συγκεκριτές αν είναι σύμφωνοι να, με την πρόταση του κυρίου Φέρχοφστάτ ή επιμένετε κύριε Σπινέλη να διεξαχθεί καταρχήν η ψηφοφορία για τη δική σας πρόταση. Θεωρώ ότι είναι μια καλή συμβιστική πρόταση του κυρίου Φέρχοφστάτ αλλά θα πρέπει να ρωτηθείτε εσείς πρώτα, πρωτίστως. Ψηφίζω για την ε, δική μας πρόταση. Um Όχι. Ωραία λοιπόν. Τότε παρακαλώ να δείξετε κατανόηση. Θα πρέπει να διεξαχθεί καταρχήν η ψηφοφορία για την ε, τροπολογία της κυρίας ε, Σπινέλη. Δεν έχω καμία άλλη ε, επιλογή. Η κυρία Χάρμς, παρακαλώ. Ε, ε, ε, θεωρώ ότι είμαστε σε μια κάπως δυσχερή κατάσταση όσον αφορά την ψηφοφορία. Σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία, κατά τις δύο τελευταίες μου επισκέψεις στην Πολωνία που συζητήσαμε για την κατάσταση εκεί, με πολύ διαφορετικές ομάδες, πανεπιστημιακούς, βουλευτές, με συντηρητικούς, προδευτικούς κλπ. Η δική μου εντύπωση ήταν ότι φυσικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον ε, για το πώς διαμορφώνεται η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο υπάρχει και ένα... Βεβαίως ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι φιλοευρωπαϊστές στην Πολωνία ε, δεν θέλουν ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πέσει σε αντιπαραθέσεις όσον αφορά την ημερομηνία της ε, ψηφοφορίας. Και επειδή εγώ είμαι υπέρ αυτής της ε, δημοκρατικής κίνησης στην Πολωνία που έχω την εντύπωση ότι παλεύουν ακριβώς για την Ευρώπη, για τα θεμελιώδη δικαιώματα και θεωρώ ότι αυτή η υποστήριξη είναι ιδιαίτερα σημαντική προς αυτές τις πραγματικές δυνάμεις στην Πολωνία, ε, θα ήθελα να μείνουμε ενωμένοι εδώ στο σώμα αυτό Ξέρω ότι δεν θα σας πείσει ιδιαίτερα κύριε Βέμπερ αυτή η πρόταση ούτε τη δική σας ομάδας και πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε το Σεπτέμβριο ε, ε, για, τον, για το Σεπτέμβριο γιατί τότε θα είναι θετικό και για μας και για την Πολωνία. Ο κύριος Βέμπερ, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το οποίο διακυβεύθηκε ε, την περασμένη εβδομάδα ήταν, ε, αφορούσε το περιεχόμενο. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους και αν συζητήσουμε επί της ουσίας ε, και αφήσουμε την ε, Κομισιόν ε, να κάνει τις εργασίες της και επανέλθουμε τον Σεπτέμβριο εμείς θεωρώ ότι εξυπηρετούμε περισσότερο την υπόθεση της Πολωνίας. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι η δική μου ομάδα συμπαρατάσσεται με την πρόταση του κυρίου Φέρχοφστατ. Ωραία λοιπόν, αλλά ρώτησα την κυρία Σπινέλη, η οποία επιμένει να γίνει η ψηφοφορία και μάλιστα ονομαστικά. Γι' αυτό δεν έχω καμία άλλη δυνατότητα από το να ε, κάνω τώρα την ψηφοφορία για την πρόταση της Ενωτικής Αριστεράς ε, όσον αφορά το σημείο αυτό να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της Τρίτης. Ζητήθηκε λοιπόν ονομαστική ψηφοφορία. Όποιος συμφωνεί όχι, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος, άρχεται η ψηφοφορία. Ε, ψηφίσατε όλοι. Ολοκληρώνεται, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τώρα έχω την πρώτη του κ. Χαφστάτ για διάσκεψη των Προέδρων την Πέμπτη, ε, στη διάσκεψη των Προέδρων την Πέμπτη να συμπεριληφθεί ε, το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια ΕΠΕΡ. κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι είναι, έχει εγκριθεί απολύτως ξεκάθαρα. Είναι πολύ ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Παρακαλώ. Εάν δεν έχετε τίποτα καλύτερο να κάνετε. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρα της ψηφοφορίας. Ε, το αποτέλεσμα ήταν ε, πολύ ίσα ίσα. Πολύ στενά τα περιθώρια. Mittwoch. Die SD-Fraktion beantragt eine Erklärung der. Έρθουμε ε, σε δήλωση της Επιτροπής στην πρόταση να συζητηθεί το θέμα μιας νέας πρωτοβουλίας στην ερευνητική διαδικασία και να μπει στη συνεδρίαση της Πέμπτης μετά τη δήλωση της κυρίας Μποργκερίνη για μια σφαιρική στρατηγική για την πολιτική ασφαλεία. Καταρχήν έχει το λόγο ο κύριος ε, Γκερέρο. Σάλομ, υπέρ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η πολιτική μου ομάδα φρονεί ότι υπάρχουν κάποια γεγονότα που αφορούν την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή ιδίω ε, γαλλικές προτάσεις οι οποίες έκαναν την αρχή και από εκεί και πέρα είχαμε επίσημες προτάσεις του κουαρτέτου ε, που ίσως αξίζουν μία δήλωση της υπάτης εκπροσώπου για να κάνουμε και έναν απολογισμό της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε. Ε, λαμβάνοντας δε υπόψη ότι στην προηγούμενη Ολομέλεια ε, είχαμε εκπροσώπους ε, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης ε, και ε, θεωρούμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε ώστε να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις και να έχουμε ένα αίσιο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος να μιλήσει υπέρ. Ο κ. Λικιώτης παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι πολύ κρίσιμη. Ε, με αφορμή και την παρουσία εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο του Προέδρου του Ισραήλ ε, και του Προέδρου της Παριστίνης, οφείλουμε ως Ευρωκοινοβούλιο να συζητήσουμε ακριβώς και να ακούσουμε και από την Επιτροπή τη θέση της, γιατί οφείλουμε να στηρίξουμε την ειρηνευτική διαδικασία. Όσο δεν προχωράει η ειρηνευτική διαδικασία, για να τερματιστεί η κατοχή της παλαιστίνης για να ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος το οποίο να συνεπάρξει ειρηνικά δίπλα στο ισραήλ τότε η κατάσταση θα είναι κρίσιμη και ως εκ τούτου η ομάδα της ευρωπαϊκής ενωτικής αριστεράς βόρειας πράσινης αριστεράς ε, στηρίζει την πρόταση των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Ευχαριστούμε κύριε Σελικιώτη. Θέλει κάποιο να μιλήσει κατά της... Εάν όχι τότε θα διεξαχθεί ψηφοφορία. Υπέρ παρακαλώ. κατά αποχές θα πρέπει να γίνει επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Η ημερήσια διάταξη λοιπόν θα αλλάξει και ως δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης την Τετάρτη θα συμπεριληφθεί αυτό το σημείο νέες πρωτοβουλίες για την ερευνητική διαδικασία. Η ομάδα του ΕΛΚ έκανε μια πρόταση η συζήτηση για το Μπαχρέιν τελικά να αντικαταστεί από μια συζήτηση για την τρομοκρατική επίθεση στον Μπακλατές. Η κυρία Γκουαρντίνη ωστόσο απέξερε την πρόταση αυτή. Αλλά θεωρητικά θα πρέπει να σας υποβάλω το ερώτημα γιατί θα μπορούσε μια άλλη ε, πολιτική ομάδα να ενδιαφέρεται. Όχι. Ωραία λοιπόν. Τότε ε, διαμορφώνεται οριστικά το πρόγραμμα εργασία, η διάταξη. Και θα έρθω τώρα στην έκθεση της κυρίας ε, Γκαρντίνη για τις οριακές τιμές εκπομπών για, ε, απαιτήσεις που, για την έγκριση τύπου για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης που προορίζονται για μη οδικά κινητά μηχανήματα.